Μετά από αυτή τη συναρπαστική και ενδιαφέρουσα ομιλία έχουμε ε, ακόμα να διεκπαιρεώσουμε την καθημερινή μας δουλειά εδώ, τρεις ακόμα επεξηγήσεις ψήφων και αρχίζουμε με την έκθεση Κοτσολίνο. και έχω την κυρία Αντρικέιν εδώ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι για το γεγονός ότι το σύνολο των ατασταλιών έχει μειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσό και ε, πραγματικά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Οι ατασταλίες στη Γεωργία συγκεκριμένα ε, περιορίστηκαν σημαντικά κατά 34%. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Ε, γιατί η Όλαφ ε, έχει αποτελεσματικό ρόλο και βοηθάει ως βασικός παράγον τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Χαίρομαι για το ψήφισμα που ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στη φορολογία επίση. Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για το γεγονός ότι οι απάτες αυξάνονται στα νέα κράτη-μέλη, κυρίως Ρουμανία και Βουλγαρία. Στους 10 της Ένωσης, τα ε, νέα μέλη ε, αυξήθηκαν κατά 8% ενώ σε αυτά τα δύο τελευταία Βουλγαρία και Ρουμανία κατά 152%. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί εκείνη η διοικητική μηχανή που να επιτρέπει με διαφάνεια να ελέγχονται οι δημόσιες προμήθειες σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Thank you. else to... Ευχαριστώ. Άλλος για την έκθεση Κοτσολίνο. Αν όχι, προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι οι μαζικές Ε, Α, όχι, συγγνώμη. Η έκθεση του κυρίου Ντόιτς και πάλι κυρία Αντρικέιν. Ε, πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Ντόιτς για την εξαιρετική του έκθεση. Η σημερινή ουσιαστική συζήτηση και το ψήφισμά μας το οποίο υπερψήφισα, είναι ε, εξαιρετική αφετηρία για τις μελλοντικέ δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική για το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα και πάλι να απευθύνω έκκληση στις κυβερνήσεις να δώσουν ε, μεγαλύτερες δυνατότητες δανειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδιαίτερα προς χώρες ανατολικές που χρειάζονται πάρα πολύ επενδύσεις και δάνεια και έχουν πληγεί τα μάλα από την κρίση επίσης. Θα πρέπει οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας και η δανειοδοτική πολιτική της ε, ΕΤΕ να συνάδουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κανείς άλλος για την έκθεση αυτή. Deutsch. Όχι. Καλώς. Και το τελευταίο τώρα επεξήγηση ψήφου αφορά τις μαζικές θηριωδίες του Τζος τη Νιγηρίας. Και πάλι κυρία Αντρικένε. Τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο γίναμε μάρτυρες μαζικών θηριωδιών στην Νιγηρία, στο Τζος. Γυναίκες και παιδιά, εκατοντάδες ε, θανατώθηκαν. Και τι χρειάζεται στην Νιγηρία τώρα, συμφιλίωση και ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των μουσουλμάνων που ζουν στο βορρά και των χριστιανών που ζουν στο νότο της χώρας. Δεύτερο, ε, η Νιγηρία ξέρουμε ότι παρά το γεγονό ότι είναι από τι μεγαλύτερε πετρελοπαραγωγέ χώρε, ο περισσότερο πληθυσμό ζει κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια και δεν επωφελείται από τη συνολική ε, ανάπτυξη. Είναι διαδεδομένη η διαφθορά ευρύτατα και θα πρέπει οπωσδήποτε και σοβαρά να αντιμετωπιστεί και αποτελεσματικά. Και τρίτον, η ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ιγυρία θα πρέπει να απευθύνεται και να ασχολείται με τα πιο σημαντικά προβλήματα και πιο ευαίσθητα θέματα για να έχουμε ε, κάποια στοιχειώδη ορατή πρόοδο, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Ο κύριος Μπέλντερ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα τελευταία νέα που ακούμε από τους χριστιανούς του ΖΟΣ είναι πάρα πολύ ανισχυτικά και μας έχουν θορυβήσει. Σε διάφορα μέρη αυτής της πολιτείας της Νιγηρίας τις τελευταίες εβδομάδες ε, χριστιανοί ε, ε, ομόθρησκοί μας ε, θανατώνονται. Στις 24 Απριλίου ε, σκότωσαν νεαροί μουσουλμάνοι, μέλη ε, μιας ένωσης, δύο χριστιανούς και μάλιστα ε, τους εξωθούν και σε τέτοιες πράξεις ατιμωρητοί σε εκρήξεις βίας και υποκινούν τα μίση και τα πάθη. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί από τις αρχές του έτους στο ΖΟΣ. Συστηματική δίωξη λοιπόν αλλοφεθρίσκων ε, παρατηρείται στην Ιγυρία. Θα πρέπει να το ξέρουν αυτά τα θεσμικά όργανα και ε, μία από τις εξηγήσει και σημαντική είναι ακριβώς οι εξτρεμιστές αυτοί οι μουσουλμάνοι από τον Ισλαμικό Βορρά εις βάρος του χριστιανικού Νότου. Κρίμα που αυτό δεν το βλέπει ε, η ε, παράγραφος 5 του ψηφίσματος. Χρειάζεται να τα πούμε αυτά με τρόπο πιο στεναρό και να το τονίζουμε. Και το ψήφισμα στρέφεται κατά ε, και παραθέτω απλουστευτικών δηλώσεων κατά κάποιον. Ναι, αλλά οι Νιγηριανοί, οι Χριστιανοί όμω υποφέρουν. Αυτά που λουστευτικά είναι αυτά που εμείς ε, σκεφτόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο, όχι όσα λέγουν ορισμένοι που έχουν δίκιο και δεν του βοηθάμε καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Νομίζω ότι είναι φρικιαστικό μια χώρα που είναι τόσο με ε, κοντινή μα όπως η Νιγηρία να γίνονται τέτοιες ε, φρικαλαιότητε. Θα πρέπει να λυθεί το θέμα μέσω του διαλόγου. Διάλογο και πάλι διάλογο και μέσω της παιδείας. Παιδεία, παιδεία, παιδεία. Ώστε να μπορέσει να επέλθει η ειρήνη στη χώρα.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 Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτή. Τα πρακτικά